Θα θυμάστε ποιες υπήρχαν πρώτα απ' όλα οι δύο προτάσεις Επιτροπής το Μάρτιο του 2009, ετής του προγράμματος της Χάγης και σύμφωνα με τις αλλαγές μετά από την ε, εφαρμογή του και εκτιμένου του Σάγκερ και τον θεσμικό ρόλο ο οποίος θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και οι προτάσεις αυτές βασίζονταν σύμφωνα με την σχετική απόφαση στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα. Τον Οκτώβριο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε αυτές τις δύο προτάσεις και ζήτησε να εγκριθεί όλη η διαδικασία στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Και εμείς είπαμε ότι θα περιμένουμε μέχρι τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαγόνης για να αναλύσουμε σε ποιο μέτρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία έγκρισης. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν και η Τσεχή και οι Σουηδικοί Προεδρία. Είπαν θα πρέπει να περιμένουμε τέσσερι σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα πριν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Βεβαίω τώρα η συνθήκη τη Λισαβόνα τέθηκε σε ισχύ. Η πρόταση για τον τρίτο πυλώνα έχει περιχειωθεί όσον αφορά την πρόταση για τον πρώτο πυλώνα. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή είπε ότι το άρθρο 74 θα πρέπει να είναι η κατάλληλη νομική βάση Βεβαίως μετά από περαιτέρω αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν το 2010 και η Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου ενέκρινε αναθεωρημένη πρόταση λαμβάνοντας υπόψη την θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν τα κράτη-μέλη. Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί ο παρόν μηχανισμός τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της ομάδας αξιολόγησης του Σέγγεν ε, έγιναν προτάσεις για να γίνει πιο αποδοτικός όλος ο μηχανισμός και η παρούσα πρόταση λαμβάνει όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τις εξελίξεις υπόψη. Επίσης, ο στόχος απ' την άλλη είναι να υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κεκτημένο Σέγγεν. Προσπάθησε η Επιτροπή να κάνει το μηχανισμό πιο αποδοτικό ε, παρακολουθώντας το πρόγραμμα, ακόμη και τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα και προσπαθεί να κάνει και επαλήθευση του, ε, της αξιολόγησης κινδύνου, ε, την ε, πραγματομοσύνη εκ μέρους διαφόρων εμπειρογνώμων. Προσπαθεί επίσης να κάνει ε, αναφορές σαφείς για να ξέρουμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται οι διάφορες συστάσεις. Και είπατε, επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ιδέουσα διαφάνεια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να μπω λίγο σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη νομική βάση. Ήδη ανέφερα ότι η του 2009 βασίστηκε στο άρθρο 66 της συνθήκης και 74 θα ήταν το διάδοχο άρθρο. Το εξετάσαμε το πολύ προσεκτικά και είδαμε ότι ίσως το άρθρο 74 είναι πολύ περιορισμένες εμβέλειες διότι αναφέρεται σε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, αλλά η πρόταση αυτή εδώ συμπεριλαμβάνει και τους διάφορους οργανισμούς. Άρα ξεπερνάει τις αρμοδιότητες του άρθρου 4. Σαν αφορά τη σωστή εφαρμογή του κεκτημένου και την πρόταση προβλέπονται κάποιες ε, επισκέψεις χωρίς να έχουν αναγγελθεί, πράγμα το οποίο ξεπερνά την ε, συνήθη διαδικασία διοικητικής συνεργασίας. Επίσης, το άρθρο 74 προβλέπεται μόνο διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αφού σκεφτήκαμε λοιπόν τη νομική βάση, καταλήξαμε στα εξή ερωτήματα. Τι κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να επαληθεύσουμε τη σωστή εφαρμοσμένη του κεκτημένου που μας επιτρέπει να έχουμε ε, έναν ε, χώρο χωρίς εσωτερικούς ελέγχους. Και θα πρέπει να έχουμε τα συνοδευτικά μέσα, τα κατάλληλα που να μας επιτρέπουν να το κατορθώσουμε αυτό. δεν πρόκειται για αλλαγή της νομοθεσίας επί της ουσίας, δηλαδή δεν αλλάγουμε, να αλλάζουμε τον κώδικα των συνόρων του Σέγγεν, αλλά δημιουργούμε ένα μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τον έλεγχο στην ε, χώρο των εσωτερικών συνόρων και να εξασφαλίσουμε ότι όταν διαβαίνουν τα εσωτερικά σύνορα δεν θα γίνεται έλεγχος στα διάφορα άτομα. Συνεχίζουμε. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει να ε, υιοθετήσουν μέτρα ώστε τέτοιου είδους εσωτερική Ελέγχη να μην είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση αυτή μπορεί να εγκριθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Ένα άλλο θέμα για το οποίο δεν βασιζόμαστε στο άρθρο 74 της συνθήκης είναι διότι έχουμε στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας ένα νέο άρθρο που προβλέπει και την αξιολόγηση των πολιτικών ε, ε, σε θέματα δικαιοσύνης ο μηχανισμός έτσι όπως προβλέπεται και η απαλήθευση για την σωστή εφαρμογή του κεκτημένου δεν μπορούν να βασίζονται σε μια διάταξη που προβλέπει μόνο συνεργασία της Κομισιόν. Και ακόμη πιο σημαντικό για σας είναι το ότι στο άρθρο 4 προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά ενημερώνονται μόνο. Πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι συνέταξαν τη συνθήκη της Λισαβόνας και έδωσαν τον ρόλο του νομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο σε θέματα ε, εσωτερικής ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν θέλουν να περιορίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουν να δοθεί σωστή ερμηνεία σε θέματα μηχανισμού αξιολόγησης του κεκτημένου του Σέγγεν. Γι' αυτό στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης, ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται αφού έχουν αρθεί οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο, αν επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο μηχανισμό για να κάνει αξιολόγηση της άρσης του ελέγχου, των ιστορικών ελέγχων, αφού όμως ε, θεθεί σε ισχύ ο παρόν κανονισμός. Άρα εδώ πέρα έχουμε ε, πρόβλημα επικάλυψης όσον αφορά την περίπτωση που προχώρησε στο Σέγγε Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στους ε, φορείς αυτού του νέου μηχανισμού που πρέπει να αντικατοπτρίζει τη θεσμική πραγματικότητα. Τα κράτη-μέλη και η Κομισιό συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη και όχι μόνο η Κομισιό με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να συμμετέχουν πλήρως στην όλη διαδικασία τα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι αυτό συνάδει με αυτό το οποίο είπαμε περί αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Όσον αφορά το δικό σας ρόλο, εκτός από την έγκριση με συναπόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει τις συστάσεις της αξιολόγησης και αν υπάρχουν ε, μεγάλες ελλείψεις θα ενημερώνεται όπως και το Συμβούλιο, αλλά τελευταίο και όχι λιγότερο σημαντικό θα γίνεται αιτήσια αναφορά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μηχανισμό αυτό. Για να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το στόχο του μηχανισμού όσον αφορά την εκτιμένο του Σέγγεν, θα πρέπει να πω ότι αν ήδη υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός όπως αυτός που αφορά τα πυροβόλα όπλα, δεν θα χρειάζεται να γίνει τέτοιου είδους επαλήθευση ώστε να μην, και η αξιολόγηση ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Ένα από τα κύρια σημεία κατά την άποψή μας είναι η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο θα πρέπει να επαληθεύεται στα πλαίσια της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν. Η αξιολόγηση μπορεί να συνίσταται σε επισκέψεις επιτόπου αλλά και σε ερωτηματολόγια που θα πρέπει να συμπληρώνει κάποιος και σε ε, επισκέψεις αυθόρμητες ή που έχουν προαναγγελθεί. Τα κύρια στουργία ενός πολιετούς προγράμματος, κάθε κράτος μέλος θα αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά κάθε πενταετία. Η Frontex θα παρέχει την ανάλυση κινδύνου και γιατί θα πρέπει να έχουν τη δική τους πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά την αξιολόγηση των εξωτερικών συνόρων και βάσει αυτής της ανάλυσης θα, θα καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα το οποίο θα σημαίνει επισκέψεις σε κάθε χώρο χώρα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο την οργάνωση επισκέψεων. Θέλουμε να έχουμε ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων. Ο κάθε κράτο χώρα θα πρέπει να ορίζει ποιοι εμπειρογνώμονε θα συμμετέχουν σε επισκέψει επιτόπου, αλλά θα πρέπει να έχουν και την απαραίτητη πείρα και προσόντα. Επίση, η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει τι ομάδε εμπειρογνωμόνων, του δικού τη μαζί με του εμπειρογνώμονε των κρατών μελών, καθώ και επισκέψεις μπορούν να γίνουν και με μέλη της Europort και της Eurojust για τις επισκέψεις επιτός. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η μείωση του αριθμού εμπειρογνωμόνων ε, σε 8 όταν ε, προβλέπεται η επίσκεψη και σε 6 όταν πρόκειται για αυθόρμητες επισκέψεις. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, Επίση, δύο εμπειρογνώμονε τη Επιτροπή ή από τα κράτη-μέλη που θα ηγούνται αυτών των ομάδων. Κάτι άλλο που προβλέπεται είναι η δυνατότητα να γίνει μία μη προβλεπόμενη αυθόρμητη επίσκεψη σε εσωτερικά ε, σύνορα από αξιωματούχους της Κομισιόν, διότι η Κομισιόν σκέφτηκε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ε, διακυβεύεται η εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών, αλλά η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στον ε, χώρο Σέγγεν, διότι πολλές φορές παραπονούνται κάποιοι πολίτες και στα εσωτερικά σύνορα τους γίνονται έλεγχοι. Γι' αυτό υπάρχουν αυτή η δυνατότητα να γίνονται αυθόρμητες μη προαναγγελθήσεις επισκέψεις. Κάποιο άλλο σημαντικό θέμα είναι βάσει το άρθρο 39 η έκθεση αξιολόγησης την οποία θα πρέπει να κάνει ο επιτόπου ε, εμπειρογνώμων και μετά στα κράτη-μέλη θα υποβάλλεται η έκθεση αυτή για να υποβάλουν ερωτήματα. Η αξιολογούμενη χώρα επίσης μπορεί να κάνει και τη δική της αξιολόγηση της έκθεσης και οι συστάσεις επίσης θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσεως στο οποίο θα προβλέπετε το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που θέλει να θέσει εφαρμογή για να διορθωθούν και κάποιες αδυναμίες. Όσον αφορά τις ε, επισκέψεις που προβλέπονται εκ των προτέρων ή όχι και τις εκθέσεις θα πρέπει επίσης να προβλέπονται κάποιες συστάσεις. Αν υπάρχουν αδυναμίες ή ελλείψεις θα πρέπει να κάνει αναφορά η Επιτροπή στο συντομότερο δυνατό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Προς το παρόν. Γίνεται επίσης αναφορά στην επιτροπολογία. Αλλά θα υπάρξει και αναθεώρη του όλου συστήματο πάνω το άρθρο 291 της Συνθήκης Λισαβόνα. Επίσης αναφέρεται η διαφάνεια όσον αφορά την διαβίβαση των συστάσεων της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, καθώς και αιτήσια αναφορά της ε, ε, αξιολογήσεις. Τελικά προβλέπεται ο μηχανισμός ε, θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που έχουν αρθεί οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Ελπίζω ότι σύντομα σας εξέθεσα την όλη κατάσταση και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Κάρλος Κοέλιο θα σχολιάσει πρωτού να ξεκινήσουμε την ε, γενική συζήτηση. Ο κύριος Κοέλιο σαν εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Οκτωβρίου του 2009 ακολούθησε τη συμβολή μου και απέρριψε την πρωτοβολία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι το πρότυπο αξιολόγηση δεν ήταν ό,τι καλύτερο και διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην συναπόφαση. Άλλαξε η νομική βάση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τώρα μία πρόταση που έχει μια νέα νομική βάση και επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην διαδικασία συναποφθήνης. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής, διότι ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να χαιρετήσω ε, την δέσμευση που είχε αναλάβει με εμά η κυρία Σεσίλια Μάστρομ. Ε, σε εξήγησε ήδη την πρώτη φορά ποιος είναι ο μηχανισμός ε, αξιολόγησης που εξήγησε η Κομισιό. Βάση επισκέψεων που γίνονται επί τόπου και έρευνες. Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να έχουν ήδη προαναγγελθεί ή να είναι αυθόρμητες. Προβλέπονται από το ετήσιο σχέδιο, δηλαδή κάθε πέντε χρόνια όλα μία φορά κάθε πέντε χρόνια όλα τα κράτη-μέλη που είναι μέλη του Σέγγεν θα αξιολογούνται και προβλέπεται και μία διασύνδεση με τη Frontex. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν οργανισμό με την εντολή της Frontex, είναι απόλυτα λογικό ο οργανισμός αυτός να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης. Επίσης, Κατά την άποψή μου υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ακόμη για μένα δεν είναι απολύτως σαφή. Δηλαδή, γιατί κάνει διαφοροποίηση η Κομισιόν μεταξύ του συστήματος αξιολόγησης που θα πρέπει να αφορά τα κράτη που είναι ήδη μέλη της Σέγγεν και του συστήματος αξιολόγησης που αφορά τα κράτη, τα υποψήφια για το σύστημα Schengen. Στο παρελθόν αυτό το είχα επικρίνει, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο επίπεδο συμμόρφωσης με τους κανόνες και από εμά. Ό,τι ζητούμε να κάνουν δηλαδή οι χώρε υποψήφιε, θα πρέπει να απαιτήσουμε να το κάνουν και οι χώρε που είναι εντό του συστήματο Σέγγεν. Βεβαίω, το άρθρο 20, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την δυνατότητα για το Συμβούλιο να εφαρμόσει ένα νέο μηχανισμό για τις νέες υποψήφιες χώρες. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είχε προβλεφθεί ευθύ εξ αρχή κάτι τέτοιο. Αν είναι ε, αναπαραίτητη μία απόφαση ενό θεσμικού οργάνου του Συμβουλίου, γιατί αυτή η απόφαση αυτή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι μιλάμε εδώ για τη διαδικασία της συναπόφαση. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη όσον αφορά αυτά τα οποία προτείνεται στο άρθρο 13 και αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και λέει όχι μόνο το Συμβολίο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται εάν ε, μία επίσκεψη αξιολόγησης ε, διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και επίσης το άρθρο 17 όπου έχει πρόσβαση το Κοινοβούλιο σε συστάσεις που έκανε το Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο μετά από μία επίσκεψη. Επιτρέψτε μου να πω κύριε Πρόεδρο ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είχε ενδιασμού το, Ευρωπαϊ... το Συμβούλιο όσον αφορά την ε, άρνηση να συμπεριληφθούν στο Σέγγεν η Ρουμανία και η Βουλγαρία χωρίς να μας εξηγεί τα στοιχεία τα σχετικά. Τι συμβαίνει με αυτή τη διαδικασία, δεν καταλαβαίνουμε τη στάση του Συμβουλίου. Συμφωνώ ότι θα πρέπει βεβαίω να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού και η Frontex και θα πρέπει να δούμε σε ποιο μέτρο εμείς πρέπει και μπορούμε να επιτρέψουμε να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία Frontex στα πλαίσια των μέσων που διαθέτουμε. Δεν ξέρω αν έχει τα κατάλληλα μέσα και το κατάλληλο προσωπικό Frontex για να κάνει τέτοιου είδους επισκέψεις. Τελικά κύριε Πρόεδρε, στερεώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Στο άρθρο 12 η Επιτροπή προβλέπει ένα σύστημα επαλήθευσης ελεύθερης διακίνησης των ατόμων. Δηλαδή, εννοεί η Κομισιό ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του εάν ναι ή όχι εφαρμόζεται σωστά ο κώδικας της Frontex. Ίσως να υπάρχουν κάποιο είδους νομικές αμφιβολίες όσον αφορά το αν αυτό το νομικό ε, έγγραφο εφαρμόζει στο σταθέρο τη, όμω την ε, Κομισιό το εξή. Γιατί προβλέπει ότι μόνο σε αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν αποκλειστικά μόνον αξιωματούχοι της Κομισιόν χωρίς ε, να προβλέπεται συμμετοχή κάποιων ε, εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη. Έτσι όπως βλέπει το σύστημα αξιωμολόγησης του Σέγγεν θεωρώ ότι είναι ένα σύστημα στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θέλουμε ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης, αλλά θα πρέπει εδώ να έχουμε και συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διότι εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν, αν δεν υπάρχει ε, έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατών μελών να μιλούμε για σύστημα αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα πρέπει, νομίζω λοιπόν, ότι αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το διασφαλίσουμε σε όλο τον μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουέλιο. Τώρα αρχίζει η ώρα των, ε, ο των συζητήσεων. Παρακαλώ τους συναδέλφους θέλουν να λάβουν το λόγο. Αρχίζοντας με τον κύριο Μπουσούτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον ε, Κάρλος ε, για την ε, παρουσίασή του. Ως εισηγητής του θέματος της Frontex θα ήθελα να έχω περαιτέρω διευκρινήσεις που αφορούν στο ρόλο της Frontex. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προτιθέμεθα να επανεξετάσουμε την πράξη σύστασης ε, αυτού του φορέα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αξιολογηθεί η Frontex. Θα ήθελα λοιπόν έτσι από την Κομισιόν ε, να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα το ρόλο της Frontex. Αν κατάλαβα καλά, ο ρόλος της ε, Frontex περιορίζεται στο να προσφέρει μια ανάλυση κινδύνου και με βάση αυτή την ανάλυση μπορούν να λειτουργήσουν ε, άλλοι φορείς ε, που ε, διεξάγουν επιτόπου επισκέψεις. Και ερωτώ, η Κομισιόν προβλέπει η Frontex να έχει και άλλο περαιτέρω ρόλο. Μάλιστα να είναι εκείνη που θα κάνει μόνη της τις αξιολογήσεις. Γιατί αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εντολή προς την Forex και προς, κυρίως να συμπεριληφθεί στο φάκελο που εξετάζουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί και σε επιπρόσθετους πόρους προς την Frontex, αν επιθυμούμε η Frontex ε, να συμμετέχει περισσότερο σε ένα τόσο σημαντικό καθήκον, όπως είναι η αξιολόγηση της ε, ικανότητας ενός κράτους μέλους να προστατεύει τα εξωτερικά του σύνορα, ακριβώς όπως προβλέπεται στο ε, κεκτημένο Σέγγεν. Θα ήθελα λοιπόν η δυνατόν η Κομισιό να μου δώσει μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Ένσιου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής Όντω χρειαζόμαστε μία αξιολόγηση του μηχανισμού του κεκτημένου Σέγγεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουέλιο για την ε, πολύ σαφή παρουσίαση του θέματος μας. Πράγμα το οποίο είναι σύνηθες στις εκθέσεις του. Και γι' αυτό μεταξύ μας τον ε, ονομάζουμε και κύριο Σέγγεν, τον συνάδελφο Κουέλιο. Θα ήθελα να πω τώρα το εξής. αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την αξιολόγηση του κεκτημένου Σέγγεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' τη μια έχουμε τις χώρες που ήδη ανήκουν στη Σέγγεν και απ' την άλλη τις υποψήφιες χώρες στη Συμφωνίας Σέγγεν. Τα κράτη-μέλη που δεν βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να έχουν κάποιο πρόβλημα διαχείρισης των εσωτερικών και εξωτερικών του συνόρων, αλλά από την άλλη πρέπει να πω ότι υπάρχουν υποψήφια κράτη-μέλη, σαν τη Ρουμανία, που παρά το γεγονός ότι σέβονται πλήρως τις διατάξεις Σέγγεν, δεν έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη του κλαμπ Σέγγεν. Θεωρώ λοιπόν ότι γι' αυτό σήμερα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή το εξής. Αυτή την άποψη δεν θεωρείτε ότι η πρόταση κανονισμού παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις συνεχίζει να προβλέπει δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις χώρες που είναι ήδη μέλος του Σέγγεν και τις υποψήφιες χώρες. Αν δεν υπάρχει κοινός μηχανισμός αξιολόγησης, πάντα θα καταλήγουμε σε διακρίσεις κατά κρατών όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι ο Κουέλιο και πάλι ανταποκρίθηκε στην σχετικά, πρόκληση σχετικά με το Σέγγεν και τον συγχαίρω για την αξιοπιστία της ε, κρίσεώς του και ε, για την επιμέλεια του. Συμφωνώ μαζί του ότι Πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της αξιολόγησης πριν την προσχώρηση και μετά όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν διότι δεν μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε την εφαρμογή του κεκτημένου εάν δεν γνωρίζετε τις ε, αδυναμίες πρώτης προσχωρήσεως στο Σέγγεν και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο επιχείρημα. Εάν δηλαδή δεχτείτε ότι υπάρχει μία δικαίωση τότε δεν θα έχει κανείς πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα πρώτης προσχωρήσεως για να γίνει μία αξιολόγηση ε, προενταξιακά διότι όπως ε, είπε ο κύριος Ράιτ θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όπως και στις συμφωνίες SWIFT. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μέτρο έναντι του οποίου να το συγκρίνουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, την τη συμμόρφωση ή όχι. Οπότε ε, πρέπει να δούμε τι συμφωνίες υπάρχουν και να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα για να δούμε ποιος είναι ο μηχανισμός αξιολογήσεως πριν από την προσχώρηση για να έχουμε ένα στοιχείο έναντι του οποίου να προβούμε σε μία σύγκριση. Επίσης όσον αφορά το, το εύρος και την αξία της αξιολογήσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην προστασία δεδομένων και νομίζω ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στα ε, βασικά δικαιώματα. Ε, ίσως δεν διάβασα καλά το έγγραφο αλλά πιστεύω ότι ε, ένα από τα προβλήματα στην παρακολούθηση, στην αξιολόγηση των κρατών μελών άπαξ και προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Σέγγεν είναι ότι όποτε γίνεται αυτή η αξιολόγηση είναι ε, περιορισμένη και τεχνική ενώ θα έπρεπε να γίνεται μία αξιολόγηση των κρατών ε, μελών από θέματα εσωτερικών υποθέσεων και ε, να δούμε αν ε, γίνεται σωστή παρακολούθηση της δημοσίας διέκησης της ε, διαφθοράς, σωστή εφαρμογή των συμπεφωνημένων κανόνων, εάν υπάρχει δίσδυση σοβαρών εγκληματιών και ούτω καθεξής, δηλαδή στοιχεία τα οποία επηρεάζουν και μειώνουν την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Βεβαίως υπάρχουν όρια στον τεχνικό χαρακτήρα της αξιολόγησης αυτής, αλλά πρέπει να δούμε ποια στοιχεία θα λάβουμε υπόψη. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω και ε, έχω κάποιο ε, ε, κάποιο προσωπικό συμφέρον όντας Βρετανή χωρίς όμως να μιλώ ε, για την υπερκυβέρνηση είναι να δούμε πόσο μπορούμε να έχουμε πρόβαση στα συστήματα παρακολουθήσεως δηλαδή όντως υπάρχει μία εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένα στοιχεία του μηχανισμού αξιολογήσεως, οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορούμε να αποκλείσουμε τελείως την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το θέμα αυτό με τη μορφή αυτή που έχει η πρόταση. Είμαι ίσως αφελής ε, και ξέρω ότι τα μη κράτη-μέλη ε, ε, φέρονται επιλεκτικά και εφαρμόζουν επιλεκτικά το Σέγγεν αλλά είμαι ειδική από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου και ευρωβουλευτών ε, στην παρακολούθηση του Σέγγεν παρόλο που δεν θέλω να το τονίσω υπερβολικά απλώ θα ήθελα να ξέρω εάν ε, το Σέγγεν έχει πρόσβαση στο ΣΥΣ δηλαδή στα συστήματα εποπτείας και παρακολουθήσεως και ε, πόσο μπορεί να παρέμβει στην εφαρμογή του Σέγγεν στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αυτά τα θέματα αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Στένοκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Κόλιο, που έκανε αυτή τη μελέτη ξεκίνησε το 2009 όταν λάβαμε τη σχετική απόφαση και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η ιδέα του αυτή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι συμμετέχουμε περισσότερο στη διαδικασία Πάντως ε, το ερώτημα που υποβάλλουμε στην Κομισιόν, το κύριο ερώτημα αφορά στην προστασία των δεδομένων. Κατά πόσον στην εντολή περιλαμβάνεται ε, και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αυτό το μηχανισμό που θα συσταθεί. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας θέση και βεβαίως ε, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον κύριο Κόελιο όσον αφορά την προσέγγιση του απέναντι στα μέλη και στα υποψήφια μέλη. Εγώ δυστυχώς ε, πρέπει να φύγω ε, για να πάω στην Επιτροπή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ε, πριν φύγω θα ήθελα να ευχαριστώ όλους εκείνους που έδωσαν να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Κόλλιο, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ, και εγώ εκ μέρους της ε, ε, πολιτικής μας ομάδας. Εγώ τα λέω τα πράγματα απλά, στεγνά, δεν τα λέω με φιωριτούρες. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατέδειξε ότι πρέπει να φαίνεται στα έγγραφα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη ανάμεσα σε αυτά που προστίθενται στη Συμφωνία του Σέγγεν και σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Εγώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχω τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, όπως και πολλοί στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που διερωτώνται, μα τι γίνεται τελικά, τι είδου ε, παιχνίδια υφαίνονται πρέπει να σας πω ότι ε, για το θέμα αυτό δεν συζητάμε καν ε, ε, στον τύπο στη Γερμανία. Διάβασε το Σαββατοκύριακο το θέμα έχει κλείσει. Αποφασίστηκε από το Συμβούλιο ότι δύο αυτέ οι χώρε δεν θα συμπεριληφθούν στο χώρο του Σέγγεν. Αυτό διάβασα στι εφημερίδε μα, ότι έκλεισε το θέμα. Και έχω το εξή αίσθημα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προφανώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα όμως έχουμε δύο έγγραφα που ε, κατατέθηκαν βέβαια πολύ καθυστερημένα και κατ' ουσίαν η συζήτηση που έγινε στον τύπο δεν ήταν επίκαιρη γιατί δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση. Πάντως η Κομισιόν είπε ότι το Κοινοβούλιο όχι μόνο πρέπει να ενημερώνεται αλλά και να συμμετέχει. Αυτό πρέπει να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια μιας διαδικασίας. Δεν συνέβη όμως εδώ. Και ως εκ τούτου ε, θέλω να μας πείτε με ακρίβεια τι θα γίνει τελικά με τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το θέμα της ε, αξιολόγησης και των προαναγγελθισών ή μη προαναγγελθισών επισκέψεων. Ποιος θα τις κάνει αυτές τις επισκέψεις και τελικά όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ε, προβλήματα, τι σημαίνει αυτό για μια χώρα. Πρέπει κανείς ε, να τα σκεφτεί όλα πολύ προσεκτικά, γιατί αλλιώς ε, φοβάμαι ότι θα καταστραφεί η ιδέα που διέπει όλο αυτό το οικοδόμημα το Schengen όπως σας είπα, προαναγγελτήσεις ή μη προαναγγελτήσεις επισκέψεις. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω καλά. Και κάτι τελευταίο που αφορά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Διάβασα μάλιστα ε, στις εφημερίδες ότι η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι η Ρουμανία ε, ε, θα μπορούσε να συμμετέχει λίγο, λίγο, όχι πολύ, λίγο, όχι πλήρως. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι και για αυτό το θέμα πρέπει τα πράγματα να διευκρινιστούν. Και αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για μας, τους βουλευτές, αλλά κυρίως για τους πολίτες στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η κυρία Φλότχα. Η κυρία Βερζάτ διορτώνει ο πρόεδρος. Δεν βλέπω κανένα ε, κανένα λόγο να με συγχαίρετε με την κυρία Φλότρ αλλά δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα εγώ είμαι η κυρία Βεντουχιά λοιπόν Είχα μία συγκεκριμένη ερώτηση και θα ήθελα να προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα διότι έχουμε εδώ τα προβλήματα της ελεύθερης διακίνησης των ΡΟΜ και στις χώρες της πλέον εμπλεκόμενες περιλαμβάνονται η Ουγγαρία και η Ρουμανία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πόσο θα χρησιμοποιήσει και θα ε, αντεπεξέλθει αυτού του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς μαζί θα μπορέσουμε και εδώ να εφαρμόσουμε τους ε, κανόνες γιατί για μένα η κατάσταση δεν είναι πολύ σαφής και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω πότε η έκθεση που μας έχει υποσχεθεί η κυρία Ρέντινγκ επί του θέματος θα μας δοθεί επιτέλους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε πάλι τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά ένα τελικό σχόλιο του εισηγητή. Ευχαριστώ. κυρία Χόρσχάμερ της Επιτροπής. Ε, ρωτήσατε αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο στραθμά. Δεν είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο το οποίο θα εφαρμοστεί διαφορετικά αλλά η διαδικασία προσχωρήσεως προβλέπει έναν διαφορετικό μηχανισμό και οι επιπτώσεις της προσχωρήσεως είναι διαφορετικές οπότε οι συστάσεις ε, προς τα κράτη-μέλη θα εφαρμοστούν άμεσα ε, στο δεύτερο μέρος της εντολής αλλά στο χώρο Σέγγεν υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός παρακολούθησης που πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπον ώστε να, εφαρμόσουμε όλες τις συστάσεις. Ε, αναφερθήκατε στην Ουγγρική Προεδρία γιατί όπως ξέρετε ε, το θέμα αυτό είναι της πλήρους αρμοδιότητας του Συμβουλίου. Η, σχετικά με τη Frontex ζητήσαμε σαν Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Frontex να κάνει μία ανάλυση κινδύνου σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Frontex θα κάνει τις επισκέψεις αυτές, αλλά απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τους καλέσει να συμμετάσχουν σαν παρατηρητές. Άρα δεν χρειάζονται τόσο πολλά, πολύ επιπρόσθετοι πόροι ε, τους οποίους ενδέχεται να χρειαστούμε την για την Frontex. Επίσης εσείς ε, έχουμε εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι τα μέτρα ε, τα οποία εμφαρμόζονται στους εξωτε, στα εξωτερικά ε, σύνορα, θεωρήσεις και ούτω καθεξής πρέπει να εφαρμόζονται για να έχουν κάποιο νόημα ή στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και θα θέλαμε να δούμε εάν η έλεγχοι της αστυνομίας που γίνονται στα εσωτερικά σύνορα δεν είναι ε, πέραν του αναγκαίου. Δηλαδή ε, πρέπει να δούμε αν η εσωτερική ασφάλεια εφαρμόζεται σωστά για να μην ε, βαρύνουμε υπερβολικά τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Η αξιολόγηση δεν είναι μόνο τεχνική, είναι και ποιοτική και αυτό αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 13.2 της πρότασης όπου λέγεται ότι πρέπει να αναλύσουμε τις ε, ε, ποιοτικέ και ποσοτικές ε, τακτοποιήσεις, δηλαδή να δούμε πώς τα θέματα αυτά εφαρμόζονται και ποιοτικά και ποσοτικά. Επίσης διαπιστώνουμε ότι το θέμα αυτό καλύπτεται εις ε, το ε, εκτιμώντας 11. Για την ε, νομική βάση που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαι σίγουρη ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια και ελπίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο έχω απαντήσει σε όλα τα συγκεκριμένα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Χοσχάμερ και τώρα δίνουμε το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Κουέιριο. Δύο μόνο θέματα έχω να παρουσιάσω. Αντιλαμβάνουμε τους νομικούς, τις νομικές αιτίες, αλλά δεν αντιλαμβάνουμε πόσο το σύστημα θα λειτουργήσει αν έχουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Εάν έχουμε διαφορετικά πρότυπα, ε, μεταξύ, ε, δύο μέτρα και σταθμά μεταξύ κρατών μελών και κρατών ε, υποψηφίων μπορεί να είναι τα μένη ψηλότερα και τα δε χαμηλότερα. Δηλαδή ή να δεχθούμε έναν υποψήφιο στο Σέγγεν και αφού γίνει μέλος του Σέγγεν στη δεύτερη αξιολόγηση να διαπιστώσει κανείς ότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις και άρα θα χρειαστεί να ληφθούν άλλα μέτρα, πράγμα το οποίο δεν έχει πολύ νόημα. Εάν ε, τα μέτρα είναι, ο πύχης είναι ψηλότερος, μπορεί να υπάρξει ε, μια αδικία για τους υποψηφίους, διότι και πολύ σωστά θα μας πούνε, ότι είμαστε πιο αυστηροί απέναντί τους που δεν είναι μέλη του ομίλου από ότι όσο είμαστε στα μέλη τα οποία είναι ήδη μέλη του Σένιεν. Άρα αυτό δεν έχει νόημα. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σοβαρά σε, αυτόν τον, ε, σε αυτό το θέμα. Και επιπλέον ε, το Κοινοβούλιο και η πρόσβασή του στα έγγραφα δεν μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως των περιπτώσεων και είναι κάτι που πρέπει να επιλύσουμε. Τώρα ε, το επόμενο θέμα δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση του Σένιον ακριβώς αλλά πολλοί αναφέρθηκαν στην ε, ε, έκθεση αξιολόγησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι κάτι που θα συζητηθεί την επόμενη πέμπτη το απόγευμα αλλά θέλω να πω εις τους συναδέλφους ότι δεν έχουμε λάβει κανένα επίσημο έγγραφο από το Συμβούλιο σχετικά με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και δεν έχουμε λάβει κανένα στοιχείο. Στην τελευταία συνεδρίαση είχα χαιρετήσει την ε, πρωτοβουλία του κυρίου Καπιτάνη, ο οποίος ε, είχε ε, λάβει ορισμένες σκέψεις από μία επίσημη πηγή αλλά είπα στην Επιτροπή ότι δεν ήταν το τελεσίδικο κείμενο ήταν ε, προσχέδια κειμένου που μας είχε στείλει ε, η Επιτροπή Σεβάλ την περασμένη πέμπτη από το Συμβούλιο και ακόμη και αν ήταν το τελικό κείμενο δεν μας το είχε στείλει επισήμως στο Συμβούλιο άρα κανείς δεν μπορούσε να είναι βέβαιος ότι δεν και το να αλλάξει μία σελίδα, μία παράγραφος ή ένα συμπέρασμα. Μόνο τα έγγραφα τα οποία μας απευθύνονται επισήμως από το Συμβούλιο μπορούν να θεωρηθούν επίσημα πράγμα το οποίο ο κύριος ε, Καπιτάνη σε μία, χέριση, σε μία κίνηση καλής θελήσεως έστειλε στα μέλη, έκτοτε όμως ορισμένα από αυτά άλλαξαν. Ε, ως εκ τούτου μην συγχαίρετε. Τα έγγραφα τα οποία ε, δίδονται είναι σημαντικά για να γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, δεν είναι όμως επίσημα. Και το Κοινοβούλιο δεν έχει επισήμως λάβει κανένα έγγραφο. Άρα όπως συμφώνησα την παρεσμένη εβδομάδα με τους χιώδεις συζητητές και όπως θα συζητήσουμε και την επόμενη πέμπτη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τη ε, διαδικασία του κατεπήγοντος που χρησιμοποίησαμε στο παρελθόν διότι δεν έχουμε στοιχεία. Κύριε Κοέγιο, ακούσαμε την παρουσίαση της Επιτροπής και τώρα ο κύριος Κοέγιο, εισηγητής, τόνισε πολύ την ε, ανάγκη του να συμμορφώνεται κανείς με την αίτηση η οποία έγινε και ολόκληρη η Επιτροπή ε, ε, Ελευθεριών πρέπει να πιέσει το Συμβούλιο για να μας δώσει στοιχεία και να επεκτείνει το κεκτημένο Σάιγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Θέλω λοιπόν να κάνω μία έκκληση πως την ε, Προεδρία, αν κάποιος εκπρόεδρος της Προεδρίας βρίσκεται εδώ θέλει να απαντήσει στην έκκληση αυτή. Όχι, τότε προχωράμε. Ε, θα αναμείνουμε όμως μία ικανοποιητική ε, αντίδραση του, της Προεδρίας και του Συμβουλίου. Γιατί ε, το θέμα αυτό έχει προκύψει κάθε φορά που συζητιέται το θέμα όπως συζητήθηκε και σήμερα. Τώρα προχωράμε στο επόμενο, το οποίο είναι μια γενική συζήτηση σχετικά με τα θέματα 6, 7, 8, 9 και 10 και 11 αν δεν απατώμε, το οποίο σημαίνει ότι ε, έχουμε την απαλλαγή 2009 Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τμήμα 3 Επιτροπή. Ο εισηγητής για όλα αυτά τα θέματα είναι ο κύριος Σιμών Μπουσουτήλ και όπως βλέπετε, βλέπω δεν αναφέρονται μόνο στις γνωμοδοτήσεις του κυρίου Μπουσουτήλ για την ε, απαλλαγή του Γενικού Προπολογισμού για την Επιτροπή αλλά ε, και για τους ε, πέντε οργανισμούς τους οποίους εμείς παρακολουθούμε. Άρα θα υπάρξει παρουσίαση από τον εισηγητή, μετά η Επιτροπή και δυνατότητα συζητήσεως εάν κάποιος θελήσει κάτι να πει από αυτόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται καθότι έχουμε καθυστερήσει. Καταρχήν να πω χαίρομαι πάρα πολύ που η συνάδελφός μας, η κυρία Βερονίκ Ματιό που ήταν η συγγήτρια για την απαλλαγή των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών είναι κοντά μας σήμερα γιατί νομίζω ότι θα την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όσα θα ακούσει. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτές τις ε, έξι γνωμοδοτήσεις στις αρχές του μήνα. Και είχαμε επίσης ε, κοντά μας εκπροσώπους της ε, Επιτροπής ε, και των πέντε αποκεντρωμένων υπηρεσιών που είναι το αντικείμενο των συζητήσεών μας. Αυτά που θα σας παρουσιάσω σήμερα βασίζονται σε ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στις αρχές του μήνα, κυρίως μετά από ερωτήσεις που υπέβαλα στις υπηρεσίες αυτές και στην Κομισιόν και με βάση τις απαντήσεις που μου έδωσαν. Θα εξτάσω κάθε μία από αυτές αυτές τις ε, γνωμοδοτήσεις που σας παρουσιάζω. Ε, πρώτον, όσον αφορά το τμήμα 3 της Επιτροπής, εκεί που γίνεται ε, λόγος για δαπάνες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής, εδώ θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά ε, στην εκτέλεση ε, των δεσμεύσεων στους τομείς ε, της ελευθερίας της δικαιοσύνης. Λυπάμαι όμως για το ότι οι ακυρώσεις πληρωμών ήταν αρκετά πολλές και παράλληλα ήταν πολλές και παράλληλα χαιρετίζουμε την ουσιαστική εκτέλεση του προγραμμάτων ε, που αφορούν στη ροή των μεταναστεύσεων και μπίπτουν στι αρμοδιότητές μας. Δυστυχώς το επίπεδο πληρωμών ήταν χαμηλότερο με ε, βάση αυτά που είχαν προβληθεί στο πρόγραμμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για τη διαφύλαξη των ελευθεριών. Επίσης, ε, καλούμε την Επιτροπή να δημοσιεύσει την ενδιάμεση αξιολόγηση για τα διάφορα ταμεία και τα προγράμματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες Τη της Επιτροπής μας και μάλιστα αυτό να το πράξει το συντομότερο δυνατόν. Γιατί η Κομισιόν μας είχε υποσχεθεί ότι θα το πράξει ε, μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Δεν το έπραξε όμως και επιθυμούμε, πρέπει να έχουμε αυτή την αναθεώρηση εάν πρόκειται να αρχίσουμε τη συζήτηση για την δημοσιονομική προεπτική κατά τα μέσα αυτού του έτους. Πάμε τώρα στην ε, γνωμοδότηση για την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων μόνο που θέλω να πω εδώ είναι ότι λυπούμεθα για το, τον τρόπο περισσότερο με τον οποίο ανατέθηκαν ε, συμβόλαια πλαίσιο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως το συζητήσαμε στις αρχές αυτού του μήνα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων. Όσο αφορά λοιπόν ε, στο EMC DDA εγώ λέω ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες ε, για τα ε, κονδύλια που έχουν προσημειωθεί στο προπολογισμό μας κυρίως όσον αφορά το EMC DDA. Πάμε στη Eurojust. Εκεί προτείνω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τη λυπή μας για το ότι ε, οι κενε θέσεις εξακολουθούν να είναι υψηλές στον οργανισμό αυτό ε, κατά 24% και πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας για το ότι συμβόλαια πρόσληψης ε, εξακολουθούν να ισχύουν. Μάλιστα προτείνω κύριε Πρόεδρε η Eurojust ε, να εξαλείψει τις ανομαλίες που υπάρχουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Όσον αφορά τώρα την Frontex, εδώ προτείνω να ληφθεί υπόψη το ποσοστό των ακυρώσεων ε, και των ε, μεταφορών του 2009 που ήταν υψηλό, ακυρώσεις και μεταφορές, ε, παρότι όπως σας είπα αυτά οφείλονται σε περιστολή του προϋπολογισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι η Frontex αυτή τη στιγμή ε, αναθεωρείται όπως επίσης και οι επιπτώσεις της χρηματοδότησης Frontex στον προεπολογισμό. Και τέλος, αυτή είναι η πιο σημαντική γνωμοδότηση που εξετάζει η Επιτροπή μας. Έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, ΣΕΠΟΛ. Εγώ λοιπόν προτείνω να λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν, υπήρξαν κάποιες ανομαλίες σε κάποιους διαγωνισμούς, κυρίως ε, αγοράστηκαν ε, προϊόντα από την Ακαδημία χωρίς να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτό έγινε και πάλι το 2009. Προτείνω λοιπόν να αναφέρουμε ότι λόγω της, ε, του αναθεωρημένου το ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αστυνομία ποτέ δεν κατέθεσε στην Επιτροπή ε, αναφερμένο κανονισμό ε, χρηματοδότησης. Ε, για αυτό το λόγο υπήρξαν συγκεκριμένε ανομαλίες που εντοπίστηκαν και πρέπει να πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ έρευνες και Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες προμηθειών δεν τηρήθηκαν και όπου τα συμβόλαια πρόσληψης που υπογράφηκαν ε, συμπεριλαμβάνουν και αυτά ανομαλίες. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ένα συμβόλαιο πρόσληψης ε, το οποίο ε, ήταν λανθασμένο εξακολουθεί να ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε την Ακαδημία να εξαλείψει αυτήν την ανομαλία αμελητή. Επίσης προτείνω να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών. Και φαντάζομαι κύριε Πρόεδρε θα το κρίνετε και εσείς αυτό απαράδεκτο. Επίσης προτείνω να πούμε ότι παρότι υπάρχει νέα ε, διαχείριση και νέα διοίκηση στην αστυνομία. Κατά το παρελθόν έγιναν λάθη τα οποία για το οποίο κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και πρέπει να πούμε ότι πράγματι ε, καταβάλλονται προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης στην αστυνομία, ε, προσπάθειες καταβάλλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, ε, προτείνω κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αστυνομική ε, Ακαδημία πρέπει να ε, συστήσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών ότι λόγω του ότι υπάρχουν πολλές ασυνέπειες και λάθη τα οποία έλαβαν χώρα στον προεπολογισμό της Ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια του 2009 γι' αυτό η απαλλαγή για το 2009 δεν πρέπει να χορηγηθεί. Και έτσι λοιπόν σας παρουσίασα τις έξι γνωμοδοτήσεις μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την προσοχή τους. Ευχαριστώ όμως κυρίως τη γραμματεία. Η κυρία ε, Κάλλαρς μοιάζει να είναι καταδικασμένη ε, να πρέπει να στηρίζει ε, ανελιπώς το έργο μου. Πάντως το χαρικά πάρα πολύ που συνεργάστηκα μαζί της και προσβλέπω κύριε Πρόεδρε στα σχόλια από τους συναδέλφους και από την Επιτροπή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε κύριε Πουζουτήλ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Φαντάζομαι είναι παρόν στην αίθουσα και επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Στεφανή Καρίγιον ε, από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα μετά από την παρουσίαση που έγινε που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές συζητήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα όσον αφορά την Επιτροπή. Απλώς θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή ευχαριστεί τον εισηγητή για την γενικά θετική άποψη την οποία εκφράζει στην εκθεσή του. Συμφωνούμε όντως ότι το 2009 είναι έτος το οποίο βλέπουμε να βελτιώνονται τα πράγματα σε αναφορά την ε, οικονομική διαχείριση των διαφόρων οργανισμών. Θα ήθελα επίσης να πούμε ότι διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της μελέτης των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, κυρίως όσον αφορά την παρατήρηση ότι θα πρέπει να υπάρξει η ε, ισομερής ε, διαχείριση και παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων. Επίσης η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει το Κοινοβούλιο ότι παρακολουθούμε έκου το τι τις ε, αξιολογήσεις που γίνονται στην, τις προσωρινές. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που αφορούν τους διάφορους οργανισμούς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τέσσερις από τους οργανισμούς, την Frontex, την Eurojust, την Frank και την ε, οργανισμό που ασχολείται με τα ναρκωτικά, ότι σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο, οι αιτήσιοι λογαριασμοί είναι μια πιστή εικόνα είναι κανονικές ε, το επίπεδο εκτέλεσης είναι κανονικό Οι πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές και λαμβάνουμε βεβαίως υπόψη όλες τις προτάσεις βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης και θα θέλαμε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι αποφάσεις που να λαμβάνονται με το πράγμα της λογικής. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιό. Α, σ' ακούσω τους συναδέλφους τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Άλβαρος, ο Άλβαρο πρώτα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολούσα τις εκθέσεις του κυρίου Μπουσούτιλ εκ μέρου τη ομάδα. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για την εργασία που επιτέλεψε. Συμφωνώ διότι προσπάθησε να επικεντρωθεί κυρίως στους τρόπους με τις οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα συστήματα. Για το ΣΕΠΟΛ ε, και εγώ έχω τις ίδιες απόψεις. Νομίζω ότι έγιναν συζητήσεις και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπισμού και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και θα γίνει και αυτό. Ελπίζω εγώ προσωπικά ότι Καλό θα είναι να είναι εδώ συνάδελφοι τη Επιτροπή Ελέγχου των Επρεπρισμού τη στιγμή την οποία συζητούμε εμείς την απαλλαγή του 2009 και για τις ε, επόμενες απαλλαγές εγώ είμαι υπεύθυνο για το τμήμα 3. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ποιες είναι οι εξελίξεις από το 2009 και εντεύθεν, να δούμε ποια ήταν τα προβλήματα, πώς ε, ε, εφαρμόστηκα λύσει για να διορθωθούν οι αδυναμίες και τελειώνοντας να πω ότι όντως συγχαίρω τον Σάιμον για την εξαιρετική δουλειά που επιτέλεσε. Κυρία Κέλλη. Ευχαριστώ. Και εγώ σε γενικές γραμμές συμφωνώ με ότι περιέλαβε στην έκθεσή του και ε, έχουμε διάφορες τροπολογίες σχετικά με τη γλωσσική διατύπωση. Ε, νομίζω όμως ότι υπάρχουν και μερικά γενικά θέματα σχετικά με τους, τους άλλους οργανισμούς. Αναφερόμαστε στην ε, απαλλαγή του 2009. Άρα δεν μπορούμε να περιλάβουμε πράγματα που βελτιώθηκαν το 2010, διότι κοιτάμε ένα συγκεκριμένο κράτος και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει συγχρόνως να συζητήσουμε τις βελτιώσεις και τις απαντήσεις σχετικά με τους διάφορους οργανισμούς. Θα ήθελα όμως πρώτα να το δω αφού το ελέγξει το ελεγκτικό συνέδριο και μετά να το θεωρήσω δεδομένο διότι ε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορεί κάποιος οργανισμός να είπε ότι θα βελτιώσει τα πράγματα ή ότι ε, γίνονται βελτιώσεις αλλά πρέπει ε, πρώτα να το επαληθεύσουμε και μετά να χαιρετήσουμε τη βελτίωση εφόσον εδώ μιλάμε για το 2000 2009. Αυτά έχω να πω επί του θέματος. Ευχαριστώ η κυρία Ματιό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον Σάιμον για την εξαιρετική εργασία που έκανε ε, στα, σχετικά με τους διάφορους οργανισμούς και λόγω πιέσεως χρόνου συμφωνώ με τις τοποθετήσεις του και η έκθεση και τα συμπεράσματά του που παρουσίασε προηγουμένως σχετικά με τους οργανισμούς αυτούς με βρίσκουν σύμφωνοι σχετικά με τις ΕΠΟΛ. Θα ήθελα να σας πω ότι όντως όπως ελέγχθη και από άλλους συναδέλφους εξετάζουμε την απαλλαγή του 2009. Άπαξ λοιπόν και ο διευθυντής άλλαξε το 2010 δεν επηρεάζει την απαλλαγή του 2009 άρα δεν συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι ο νέος ε, διευθυντής έχει κάνει πολλά για να βελτιώσει την κατάσταση και θα δούμε φέτος. Τώρα όμως δεν συζητάμε το 2010, συζητάμε το 2009 και την απαλλαγή του 2009. Άρα συμφωνώ με τον εισηγητή και γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με αυτή τη, αυτό τον οργανισμό και για μένα ό,τι συνέβη το 2009 δεν ήταν αρκετά καλό ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε απαλλαγή. Άπαξ όμως, να χορηγήσουμε απαλλαγή. Άπαξ όμως και είμαστε στην Επιτροπή των Ελευθεριών. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα με τον οργανισμό ΣΕΠΟΛ. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την θέση που της αρμόζει στο Governing Board εφόσον δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί προηγουμένως μιλήσαμε ε, για ιδιωτικές δαπάνες που χρησιμοποίησαν τα χρήματα των φορολογουμένων. Μιλήσαμε και για τις ε, ε, παρατυπίες του Διευθυντή ο οποίος απεχώρησε αλλά δεν νομίζω ότι ήταν στο ύψος των περιστάσεων ο Διευθυντής αυτός και δεν νομίζω ε, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ε, αντάξια της θέσεώς τους. Άρα θα έπρεπε να ξαναδούμε την ε, διάρθρωση είτε να συνδυάσουμε την ΣΕΠΟΛ με την Ευρωπόλ ή ενισχύοντας τη ΣΕΠΟΛ. Δεν πιστεύω όμως ότι ο οργανισμός αυτός παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνει αυτή τη στιγμή ο Διευθυντής δεν πιστεύω ότι μπορεί να επιβιώσει στην ισχύουσα κατάσταση και καλό θα ήταν το Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα αυτό διότι δεν είναι σωστό να διατηρούμε μια τέτοια δομή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Ορισμένα τελικά συμπεράσματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα καλά τους λόγια και να τελειώσω με τα σχόλια για την ΣΕΠΟΛ διότι θυμάστε ότι πέρυσι δεν δώσαμε στην ΣΕΠΟΛ απαλλαγή για το 2008 και η ε, Επιτροπή Προπολογισμού αποφάσισε μόνο πριν από λίγες μέρες να δώσει την απαλλαγή του 2008 πράγμα το οποίο επιζητούσαν επί τόσο καιρό. Αλλά η απαλλαγή του 2009 θα χορηγηθεί από την Ολομέλεια. Δεν μιλάμε όμως τώρα ούτε για το 2008 ούτε για το 2010 αλλά για το 2009 όπου διαπιστώνουμε ακόμη παρατυπίες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εστιαστούμε στο θέμα αυτό και δεν αμφιβάλλω ότι δεν έχουμε λόγο να μην δώσουμε ε, απαλλαγή διότι όπως μας είπε ε, η κυρία Ματιό πρέπει να σκεφτούμε ε, αν έχει λόγο να διατηρηθεί αυτή η δομή ή πρέπει να ενσωματωθεί σε μια άλλη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, όπως σωστά είπατε, θέλετε ένα ηχηρό νόμισμα. Βλέπω ότι η Επιτροπή σηκώνει το χέρι. Θέλετε κάτι να μας πείτε, μία τεχνική διευκρίνηση. Διότι η απαλλαγή από ό,τι, από κατάλαβα δεν θα δοθεί για το 2008, απλούστατα θα κλείσουν οι λογαριασμοί και δεν θα υπάρξει ποτέ απαλλαγή για το 2008. Πρέπει όμως να κλείσουμε τους λογαριασμούς για να μπορέσει να ε, λειτουργεί το επόμενο οικονομικό έτος, απλώς. Ωραία, σαφέστατο λέει ο Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι ε, την 5η 3 ε, Φεβρουαρίου στις 12 και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τώρα προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι το 12 η εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα και την θέσπιση αδείας εξαγωγής καθώς και μέτρων εξαγωγής διαμετακόσμησης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματα και πυρομαχικά. Η συγητής είναι η συνάδελφος Βερονίκ Ματιέ. Ε, ε, η Επιτροπή ε, ζήτησε να εφαρμοστεί ε, το άρθρο 50 αλλά δεν έγινε αποδεκτή η αίτηση οπότε τώρα θα ακούσουμε την ομιλία της συναδέλφου Ματιώ μετά την Επιτροπή και μετά θα γίνει συζήτηση. Η κυρία Ίντβελτ. Ε, δεν ήμουν εδώ, ίσως το είπατε, αλλά προβλέπαμε μία συνεδρίαση ε, και κλεισμένων των ε, θυρών. Θα λάβει χώρα, ναι, ναι, στις 6 θα ξεκινήσει αυτό το θέμα και ε, αν είμαστε έτοιμοι θα το πράξουμε. Λοιπόν, κυρία Ματιό, εάν μας βοηθήσετε με μία σύντομη παρουσίαση θα το εκτιμούσαμε. Κατανόησα το μήνυμα κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι. Η πρόταση κανονισμού ανταποκρίνεται στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρει το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου των, ε, του ΟΗΕ για τα πυροβόλα όπλα και θέσει άδειε εξαγωγή, καθώ και μέτρου εξαγωγή και διεντάγματα για πυροβόλα όπλα μέχρι εξαρτήματα και πυρωματικά. Αυτό γίνεται για να μπορέσουν ναι, να ελεγχθούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές τέτοιου είδου ε, πυροβόλων όπλων προς τρίτες χώρες. Η εναρμόνιση είναι καλόδεκτη. Αυτή τη στιγμή η κάθε εθνική νομοθεσία επί του θέματος διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι λοιπόν σημαντικό να υιοθετήσουμε ενιαία μέτρο ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με τα κρατών μελών και να γίνεται νόμιμα η μεταφορά όπλων. Θα πρέπει να υπογραμμίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των ΜΜΕ που είναι πάρα πολύ δυναμικές στην αγορά. Δεν θα πρέπει να έχουμε παχθεί και άχρηστη ε, ε, γραφειοκρατία που θα τις τους κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, συνθήκες ε, θεμητού και υγιού ανταγωνισμού για τις μιμιές σε σχέση με αυτές των τρίτων χωρών. Στο κείμενό της η Επιτροπή προσπάθησε όλες αυτές τις ε, απαιτήσει να τις ισοσκελίσει παρά το γεγονός ότι κάποιοι ορισμοί είναι απαρχαιωμένοι. Πώς ορίζεται το πυροβόλο όπλο η χρησιμοποίηση του μολύβου, ενώ σήμερα δεν χρησιμοποιείται πλέον για λόγους προστασίες του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι προκαλεί μολυβδίαση σε κάποια ζώα. Θα ήθελα να χαιρετήσω επίσης την διαδικασία την ε, απλοποιημένη διαδικασία εξαγωγών και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις προσωρινές εξαγωγές όπλων καθώς και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει επανεισαγωγή και εξαγωγή του όπλου για λόγους συντήρησης. Θα πρέπει οι διάφορες διαδικασίες να μην είναι χρονοβόρες και δεν θα πρέπει σε περίπτωση που ζητείτε άδεια ε, για την εξαγωγή όπλων να προβλέπεται μεγαλύτερη χρόνος από 60 ημέρες. Επίσης άλλα θέματα ε, προς θεμιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις ε, ευθυγραμμίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ματιό την παρουσίαση της εκθεσής σας. Δίνω το λόγο τώρα στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ακούσουμε την Επιτροπή. Τον κύριο Ντιντερή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή θα θέλει να ευχαριστήσει κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πρόταση και βεβαίως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κυρίως ε, την εισηγήτρια, την κυρία Ματιέ, όπως επίσης και τον κύριο Γιακολίνο που είναι παρόν και αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής εμείς παρουσιάσαμε ε, το στόχο και το εύρος αυτής της πρότασης. Η, η συγκήτρια ανέφερε ότι αυτό που απομένει είναι η επικύρωση της ε, συμφωνίας ε, ακόμα αυτή εκρεμή, Ο κανονισμός λοιπόν θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί και εσείς είπατε δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας στο ότι είναι απαραίτητο παρόλα αυτά να διασφαλίσουμε την εφαρμογή υποχρεωτικών σχεδίων και το πνεύμα του πρωτοκόλλου. Επίσης, να διασφαλίσουμε μία συνέχεια και μία συνέπεια. Η συνέπεια πρέπει να διασφαλίζεται μαζί και να είναι η συνέχεια άλλων νομοθεσιών που έχουν λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ε, θα ήθελα επίση να μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλήρως στη διάθεσή σας ε, για να σας βοηθήσει. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για το Συμβούλιο. Ε, για συγκεκριμένα θέματα τα οποία ενδεχομένως χρειάζονται κάποια διευκρίνηση. Επίσης για να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η ταχύτατη έγκριση του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ εκπρόσωπο της Επιτροπής. Τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα θέλαμε να ακούσουμε το Συμβούλιο. Κύριος Λάγιος Ράτσι από το Συμβούλιο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας μπορώ να σας πω ότι λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του φάκελο αυτό. Κάνουμε σοβαρές έρευνες. Ήδη ασχοληθήκαμε σε δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου με το θέμα αυτό και προβλέπουμε και κάποιες συμπληρωματικές συνοντήσεις για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Ο σκιώδης συζητής είναι ο κύριος Τζακολίνο. Θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση συμπληρωματική. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν παρεμβαίνω ως ε, είμαι εισηγητή στην άλλη επιτροπή που είναι και αυτή συναρμόδια, είμαι εισηγητή στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Άκουσα λοιπόν τις ε, παρατηρήσεις <clears throat> και τις ε, συστάσεις κυρίες Ματιώ, όπως άκουσα με μεγάλη προσοχή και εκείνες τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν τόσο από την Κομισιόν όσο και από το Συμβούλιο. Προφανώς λοιπόν το θέμα αυτό αφορά εμπορικές διαδικασίες ε, και κάτω από το πρίσμα της ασφάλειας. Βεβαίως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε η κυρία Ματιώ, η, η και πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια Επιτροπή ανέφερε ότι ε, κάποιες αρχές ε, σε κανονιστικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμόζονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι θα υπάρξει ε, και κάποια σωστή επιχειρηματολογία για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Οι τροπολογίες ε, νομίζω ότι μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 3 ε, Φεβρουαρίου, ενώ στην άλλη επιτροπή που είναι αρμόδια επί της ουσίας, οι τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε αυτό που είπε η κυρία Ματιέ σε σχέση με τις ημερομηνίες και τις εργάσιμες ημέρες. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το εξετάσουμε, όπως μπορούμε να εξετάσουμε και το θέμα της θέσης του κανονισμού στην αρχή η Επιτροπή είχε πει τέσσερις μήνες, ενώ τώρα η κυρία Ματιέ μιλάει για 18 μήνες. Αυτά είναι θέματα που θα μας ε, απασχολήσουν. Ε, θα απασχολήσουν τους ε, εισηγητές τόσο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, όσο και τους εισηγητές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο Η κυρία Γκόμες ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Βεγρονίκ Ματιέ για την έκθεσή της όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Όταν διάβασα την έκθεσή της πρέπει να πω ότι ανησύχησα διότι δεν γίνεται αναφορά στην ανάγκη να υπάρχει σύνοχη με την κοινή θέση που εγκρίθηκε στο τέλος της Γαλλικής Προεδρίας το 2008, κώδικα δηλαδή συμπεριφοράς, για τους κανόνες που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών των στρατιωτικών ε, ε αντικειμένων. Εδώ θα μου πείτε ότι πρόκειται για πυροβόλα όπλα που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά τα κυνηγητικά όπλα είναι τα όπλα τα οποία αποτελούν πραγματικά όπλα μαζικής καταστροφής σε κάποια άλλη πύρο, στην Αφρική Φερρυπίν. Και πολύ συχνά εμείς εξάγουμε αυτά τα μικρά όπλα ε, στις χώρες αυτές και πραγματικά χρησιμοποιούνται από τα μικρά παιδιά που στρατολογούνται ε, σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να είναι συνεκτική. Και αν έχουμε έναν κανονισμό αρκετά απαιτητικό σε θέματα ελέγχου εξαγωγών της στρατιωτικής τεχνολογίας, δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε όταν έχουμε να κάνουμε με αυτά τα όπλα, τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι το Κοινοβούλιο κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ώστε ο κώδικας συμπεριφοράς να γίνει από νομικής πλευράς δεσμευτικός. Εγώ στη χώρα μου και ξέρω ότι σίγουρα αυτό συμβαίνει και σε άλλα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Έννοιας. Πολλές έρευνες στην αστυνομία και στις στρατιωτικές αρχές που μπορούσαν όντως να δώσουν το πράσινο φως για τις εξαγωγές τέτοιου είδους όπλων, αλλά ανακάλυψα ότι πολλά όπλα εξάγονται με μια άδεια που παρέχεται από κάποιες αρχές όπλα τα οποία είπαμε ότι χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς ε, λόγους, για μη στρατιωτικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς τελικά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεκτικοί και θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η απόψή της για το θέμα αυτό και επίσης να ζητήσω από την εισηγήτρια να το εξετάσει αυτό το θέμα. Διότι νομίζω ότι συνοχή θα μας βοηθήσει σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα. Ευχαριστώ. Έχουμε, πρέπει να σας πω, γιατί για το επόμενο θέμα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες που είναι εδώ και μας περιμένουν. Περιμένω να τελειώσουμε. Παρακαλώ λοιπόν, περιοριστείτε, να είστε συνοπτικοί. Ο κύριος Ένσιου. Da, în calitate de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 Uh, nu Δεν πιστεύω ότι αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται για να γίνονται μασικέ δολοφονίες όπως ελέγχθη. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό ήθελα να πω. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να έχουμε ισορροπία μεταξύ του να σταματήσουμε την παράνομη οπλοθυρία και απ' την άλλη να προστατεύσουμε την ε, βιομηχανία που παράγει αυτά τα όπλα. Εάν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξάγουμε όπλα, σίγουρα άλλες αναδυόμενες χώρες θα πάρουν τη θέση μας και εκείνοι θα κάνουν τα στραβά μάτια σε κάποιους ελέγχους σε σχέση με το τι κάνουμε εμείς. Θα ε, ήθελα να έχω μιλήσει με την κυρία Ματιό και με την ομάδα μου για τις διάφορες απόψεις ε, της αποκλίνουσης, αλλά είμαι σίγουρη τελικά θα καταλήξουμε σε λύση. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Λοιπόν, ουσιαστικά ε, χρησιμοποιούνται τα όπλα στις σφαγές σε σχολεία και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου ε, πρέπει να προστατεύσουμε ιδίως τους πολίτες και όχι τόσο τις βιομηχανίες. Ε, θα έλεγα να εφαρμόσουμε πλήρως το άρθρο 10 και να μην διευκολύνουμε τις εξαγωγές όπλων για αναψυχή διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά γράφει για τη χρήση των όπλων στο έγγραφό της. Ε, θα ήθελα όμως μια γραπτή απάντηση ε, σε τι εννοείται όταν μιλάτε για άλλα ε, όταν εξετάζετε αυτό τον κατάλογο. Ευχαριστώ. Τώρα τελικό σχόλιο από την εισηγήτρια κυρία Ματιά Όχι, δεν χρειάζεται κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα ανακοινώνω ότι είχαμε για σήμερα το απόγευμα και το σημείο 13 σχετικά με το κατάλογο ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπει στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση ή τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση κατάρτιση αυτού του καταλόγου με εισηγείται την κυρία Τάνια Φαγιόν αλλά την ευχαριστούμε διότι ευγενώς ε, ε, συνένεσε στο να μεταφερθεί η προσυζήτηση αύριο μετά την ψηφοφορία και έτσι θα μπορέσουμε ακόμη σήμερα ε, και κλεισμένων των θυρών να συζητήσουμε το σημείο 14 σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με τις συμφωνίες PNR της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων και μία ενημέρωση σχετικά με τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων PNR από τον φιλοξενούμενό μας ε, κύριο Ράινχαρτ Πρίμπε ο οποίος θα ε, μας ενημερώσει εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω θα μπορέσουμε να έχουμε και μία σύντομη συζήτηση. Ως συνήθως πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε τους διερμηνείς μας εάν μας δώσουν λίγα με επιπρόσθετα λεπτά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην υπερβούμε το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι